Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε. Κυρίσω την ε, επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στις 23 Ιουνίου 2016 σε απόλυτη συμφωνία με τις ε, πολιτικές ομάδες συγκάλεσα αυτή την έκτακτη συνεδρίαση δυνάμει του άρθρου διακόπτει ο πρόεδρος